Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ πολύ να είστε πιο προσεκτικοί τη στιγμή που ψηφίζουμε. 2.43 υπέρ. Κατά. 2.43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ. Κατά αποχές. Και πάλι ηλεκτρονικά για την 2.44. Εγκρίνεται και μάλιστα άνετα. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.59 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 259. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίν, αποχές εγκρίνεται. 2.60 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,78 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 282 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 283 υπέρ, κατά, αποχές. Λοιπόν, τη 283 θα την κάνουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην ΤΕΒΕ 5 υπέρ κατά αποχές και εδώ ηλεκτρονικά παρακαλώ γιατί δεν είδα αρκετά χέρια να σηκώνονται είμαστε στην ΤΕΒΕ 5 ή εγώ είμαι άχρηστη και δεν σας βλέπω Θα σας βάλω έναν ένα ναι να έρθετε εδώ να δείτε τι περνάω. Ωραία, βιάζομαι. Ναι, αλλά καμιά φορά εμείς πρέπει να αλλάξουμε σελίδα όταν έχουμε τη συμβιβασμό και κοιτάμε στην πίσω σελίδα και δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι γίνεται. Δεν έχουμε το χρόνο. Καλά, θα τα λέω πιο αργά, υπόσχεται η πρόεδρος. Λοιπόν, πού ήμουνα. 2,85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.86 και 7 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 2.89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 2.93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.95 τμήματικά πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.96 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9.4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ, το δεύτερο τμήμα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και το υπόλοιπο των ΔΕΒΕ μαζί Ξεκινάμε. Α, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να τα ψηφίσουμε εν μπλοκ. Λοιπόν, δεβένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεβε 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεβε 3. Υπέρ κατά αποχές ΤΕΒΕ DV11 υπέρ κατά αποχές ΤΕΒΕ DV12 υπέρ κατά αποχές στη 12 παρακαλώ ηλεκτρονικά απορρίπτεται ΔΕΒΕ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 18 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στα εκτιμώντας. Πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έξι και οκτώ που είναι ήδη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 7, 9 και 14 ταυτόσιμες υπέρ. 7, 9 και 14 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. 11 με συγχωρείτε κατά, ε, αποχές εγκρίνεται, οι 11 και οι 12 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε τώρα στο συμβιβαστικό, πρώτη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτη συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 41 και 42 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 48 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εδώ και πάλι 40, 49 ε, ηλεκτρονικά Απροβάδα. Εγκρίνεται λοιπόν 50 σε δύο τμήματα υπέρ, το πρώτο τμήμα κατά, αποχές, σας τα λέω στα σοβαρά τώρα. Συγγνώμη, το ΕΛΚ δεν, ψηφίζει. Θα σας το πω ανοιχτά. Γιατί από εκείνη την πλευρά δεν ψηφίζει κανείς. σα το λέω απολύτως σοβαρά. Είμαστε στην 50. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέμπτη συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 σε τέσσερα τμήματα υπέρ το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 71 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβιβασμός 7 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 και 86 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίνονται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 με συγχωρείτε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σύμβασμος 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 με μια προφορική τροποποίηση που την έχετε στα χαρτιά σας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 121 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 122 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 19 υπέρ 11 εναντίον καμία αποχή συγχαρητήρια κυρία Μπεθέρα Seguimos con la votación. Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Περνάμε στην επόμενη έκθεση για τα δικαιώματα της ε, γυναίκας σας στην εταιρική σχέση με τις ανατολικές χώρες. Ξεκινάμε με την ψήφιση. Τροπολογία 15 υπέρ. αν συμφωνείτε, να καθίσετε παρακαλώ. Και ξεκινάμε με την επόμενη ψηφοφορία. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Της ε, νομικής επιτροπής 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 21, άρχεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε πάλι έλεγχο. Ψηφίζουμε την 22 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 36 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμ... Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ντροά 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 8 υπέρ να ελέγξουμε την 51 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Εγκρίθηκε 51. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δρόα 17. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δρόα 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 52. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 63 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 63 πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. 64 υπέρ. Να ελέγξουμε ποιο. Το δεύτερο τμήμα της 63. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Μάλιστα. 64 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 66 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα καταπίπτει 67 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε συμβασμός 11 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε Τοπολογία 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ντρουά 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Δρουά 3 καλύπτεται αυτή η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Δρουά όχι καλύφθηκε. Συμβιβασμό 12 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίθηκε. Τροπολογία 79 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίφθηκε. Ντρουα 5 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίθηκε. Τροπολογία 80 υπέρ κατά Απόχε. εγκρίθηκε. 81 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 83 υπέρ 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Δρά 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 85 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Δρουά 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε τροπολογία 1 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε δρούα 5 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ. Να ελέγξουμε, εντάξει, ελέγχουμε την 3. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά ποσές απορρίφθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Να ελέγξουμε ποιαν. πια να ελέγξουμε, τη 12. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που είχα πει. Μάλιστα. Σιγά σιγά τώρα τερματίζεται η υπομονή, πώς να το πω. Ahora la enmienda 12. Mm. Sí. Pasamos a la enmienda. Περνάμε στην τροπολογία 13. Αν θέλετε επίση να κάνουμε και έλεγχο τη 11. Ναι, ωραία, εντάξει, εμπρό. Ελέγχουμε την 11. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Ωραία. Πάμε στην 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα και ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. 22 ψήφοι υπέρ. 3 εναντίον και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. vamos a votar el ultimo... Λοιπόν, ψηφίσουμε την τελευταία τελική έκθεση. Κουραστήκαμε βέβαια όλοι, αλλά ολοκληρώνουμε και θα ξεκινήσουμε και με τις συζητήσεις μετά. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι δεν ήταν η καλύτερη ημέρα σήμερα για μένα με τις ψηφοφορίες των οποίων προέδρευα. Συμβασμός 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα σοβαρά, εντάξει, ελάτε. Να κάνουμε έλεγχο για το συμβασμό 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. εγκρίθηκε. Έχω ακόμα κάποιε ικανότητε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, περνάμε στην τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίθηκε. 37. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίθηκε. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίθηκε. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Το Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 42 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 43 υπέρ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε δεύτερο υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 44 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 45 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά απόχε, εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά απόχε, εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά απόχε, απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά άποχέ, εγκρίθηκε Συμβασμό 4 υπέρ κατά απόχε, εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 54 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 55 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 56 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε όχι δεν το ξέρω αυτό θα το ελέγξουμε ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή ηλεκτρονικά άρχεται Μάλιστα απορρίφθηκε λοιπόν 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε να ελέγξουμε την 58 ηλεκτρονικά εντάξει άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Απορρίφθηκε λοιπόν. Λοιπόν, το αρχικό κείμενο στην παράγραφο 2. Όχι, καταπίπτει αυτό γιατί υιοθετήθηκε άλλη τροπολογία. 59 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 61 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 68 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 68. Εντάξει. Εγκρίθηκε. 69 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Θα ψηφίσουμε την 70 τώρα. Σε 7 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Έκτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έβδομο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 72 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε 73 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε συμβασμός 5 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 79 σε τρία τμήματα πρώτο υπέρ να ελέγξουμε ποιαν. Την 78. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 78 ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. 79. Σε τρία τμήματα. Πρώτο. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 79 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Δεύτερο τμήμα της 79. Εντάξει εγκρίθηκε. Και τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Α, απο, ε, κατά απο, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 92. Ψηφίζεται. Απερίφθη. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 97 υπέρ, κατά, αποχές, δε, απορρίπτεται. 98 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 99 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή η 100 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφεται 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίο 1 υπέρ κατά αποχές α δεν βλέπω έλεγχος για την 1 ψηφίζεται απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 α όχι καταπίπτει 4 αρχικό κείμενο πίπτη και αυτό 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 με μια προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζεται. 15 υπέρ 9 κατά 2 αποχές. Καλή τύχη λοιπόν κυρία Ρενά. Uh, um, Για να συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη που είναι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωση για την Ισότητα των Φύλων. Η Κλέρ Μούντι είναι η συγγήτρια. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως και όταν μιλάμε για κονδύλια ξέρω πως οι σφιγμοί αυξάνονται ε, Τέλο πάντων δεν είμαι και σίγουρη, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να κάνω μια εισαγωγή για την έκθεση αυτή εδώ στην Επιτροπή μας. Ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, ένας, είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά ισχυρό γιατί υπάρχει για να εφαρμόζει τις προτεραιότητές μας και κυρίως για να εφαρμόζει και τις αξίες μας και σε πολλές περιπτώσεις δεν βλέπουμε να στον προϋπολογισμό να αναφέρονται τα θέματα φύλου όπως αναφέρονται στις συνθήκες και σε κάθε πολιτική που ακολουθούμε. Βρίσκεται σε συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα στο ΕΚΤ, στα δικαιώματα, στο Horizon 2020, ε, στις δαπάνες εκεί και σε άλλα προγράμματα, αλλά σε άλλους χώρους αυτό που βλέπουμε είναι να παραπέμπουν στις γενικές αρχές της ισότητας των φύλων, αλλά πολύ λίγα προγράμματα πέραν αυτών που έχουν συγκεκριμένους στόχους, που να περιγραφούν συγκεκριμένους πόρους και κονδύλια που θα διατεθούν για το θέμα της ισότητας. Όταν λοιπόν μιλάμε για σχεδιασμό και εφαρμογή, τότε δεν έχουμε ε, κάποιους δείκτες που να κάνουν αξιολόγηση των κονδυλίων, το αν υπάρχουν τα κονδύλια και το πώς χρησιμοποιούνται. Έχουμε το πολιετές ε, πλαίσιο που φτάνει μέχρι το 2020 και εκεί είχαμε κάποιες ε, πολύ ε, ισχυρές διατυπώσεις για θέματα φύλου, αλλά η στρατηγική η ίδια δεν έχει καλύψει όλες τις απαιτήσεις και νομίζω ότι δεν έγινε και καμία αναφορά στην ισότητα των φύλων στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολίτους. Η έκθεση εστιάζει σε τρεις χώρους χρηματοδότησης που θεωρούμε κομβικούς δηλαδή στα Ευρωπαϊκά Διαστατικά και Επενδυτικά Ταμεία, εξετάζουμε την πρόσβαση, για παράδειγμα, στην απασχόληση και πέραν των όσων λειτουργούν, έχουμε τονίσει και κάποια σημεία στα οποία χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει συστική, συστηματική μέθοδος για να γίνεται το mainstreaming και επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε και τι συμβαίνει ε, με τα κοινωνικά επιδοτήματα για τις κοινωνικές υποδομές, για παράδειγμα για τις υπηρεσίες φροντίδας. Επίσης τα δικαιώματα, ε, τα πολιτικά δικαιώματα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές ε, κυρίως στα, στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και στην ε, έκθεση αυτή λέμε πως έχει μειωθεί εκεί η χρηματοδότηση το 2011 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για το συγκεκριμένο αυτό. Στο 2012 φτάσαμε στα 19,5, το 2013 πήγαμε στα 18 και μέχρι το 2016 είχαμε πέσει στα 14 εκατομμύρια χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν προφανέστατα χρειάζεται να δούμε αυτή τη μείωση Επίσης θέλουμε να μας δοθεί περισσότερη σαφήνεια για άλλους κλάδους όπου έχουμε δαπάνες ε, τέτοιου είδους για την καταπολέμηση της βίας σε όλες τις διαστάσεις της και θα πρέπει να συλλέξουμε και αυτά τα στοιχεία τα οποία ανακατανέμονται κατανέμονται αναφύλο. Και μετά έχουμε την έρευνα και τεχνολογία, το τρίτο κομβικό, γιατί στο Horizon 2020 για το mainstreaming έχουμε συγκεκριμένες δράσεις και η στήριξη για τα ερευνητικά κέντρα που έχουν πολιτικές ισότητας των φύλων όντως ε, έχουν εγγραφεί και έχει γίνει κάποια προσπάθεια και με το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα, αλλά ακόμα και εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Επίσης, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για μια οπισθοδρόμηση και από χώρισε από κάποιες εξαιρετικές αρχές, για παράδειγμα με το έγγραφο για το, τις γυναίκες στην επιστήμη, ε, όπου το θέμα της ισότητας των φύλων ε, κάπως πνίγεται ανάμεσα σε έναν ευρύτερο τίτλο για θέματα ερευνητικά. Οπότε, ναι, Αναγνωρίζεται βέβαια η ισότητα των φύλων. Στην εξωτερική δράση έχουμε το σχέδιο δράση το σχετικό στη μετανάστευση και στο άσυλο και τα σχετικά ταμεία. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους ad hoc μηχανισμούς γιατί δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ε, που να θεωρείται ad hoc και όπου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Η βασική σύσταση λοιπόν είναι να χρησιμοποιείται ε, σε όλα τα επίπεδα η αξιολόγηση ε, της χρήσης ε, της ε, η αξιολόγηση του κατά πόσο βοηθά στην ισότητα των φύλων κάθε συγκεκριμένο ταμείο και να εφαρμόσουμε με μεγαλύτερη προσοχή όλα τα ωραία λόγια που έχουμε συμπεριλάβει στις κατά καιρούς δηλώσεις μας. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους δείκτες, όχι μόνο για την εφαρμογή, αλλά και στα στάδια της επιτήρησης και της αξιολόγησης και τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και τέλος χρειάζεται τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση έτσι ώστε όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή των project αυτών να γνωρίζουν ποια είναι η διάσταση φύλου που τους αφορά συγκεκριμένα στη δουλειά τους. Προφανώς είναι και ευρύς ο χώρος και μάλλον περίπλοκος. Προσπάθησα να καλύψω στην έκθεση όσο περισσότερο μπορούσα, αλλά με μεγάλη χαρά θα ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων και για τις τροπολογίες, αλλά και για την έκθεση την ίδια για να προχωρήσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στους σκιώδες ηγητές. Θα ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η μπάρμερα Ματέρα αυτή τη στιγμή είναι σε άδεια μητρότητα και αυτή είναι η σκιώδη από την πλευρά του ΕΛΚ και δεν μπορεί βέβαια να παραστεί, αλλά θα σα διαβάσω τα, τις σημειώσεις που μου έστειλε. Και σα ευχαριστώ πολύ και μια φορά ακόμα σα ζητώ συγγνώμη. Καταρχήν ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που έκανε και θα θέλαμε να κάνουμε και κάποια σχόλια σχετικά με την έκθεση αυτή. Δηλαδή στην Επιτροπή Γυναικών έχουμε δουλέψει σκληρά τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να έχουμε μια αξιολόγηση ετήσια του τι γίνεται για τα θέματα του φύλου μέσω του προπολογισμού και έχουμε καταφέρει στην διαδικασία προϋπολογισμού να συμπεριλάβουμε ε, κάποια κονδύλια ε, και κάποιες δαπάνες για να πετύχουμε την ισότητα. Και για να το καταφέρουμε αυτό και για να σεβαστούμε τις στρατηγικές μας δεσμεύσεις έχουμε πει πως πρέπει να χρηματοδοτούμε προγράμματα στα πλαίσια των πιο βασικών ε, γραμμών του προπολογισμού, δηλαδή το κοινωνικό ταμείο, ε, το, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως επίσης και στα διαρθρωτικά και τα επενδυτικά ταμεία. Να σας πω προς τα πόλα πως το mainstreaming θα πρέπει να θεωρείται μια εναλλακτική λύση, ε, διαφορετικά θα πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για όλες τις πολιτικές για το θέμα του φύλου. Και επίσης θα πρέπει στα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαφορετικά Ταμεία να ενισχύσουμε τη διάσταση αυτή, γιατί μέσω αυτού του ταμείου θα πρέπει να εφαρμόζουμε ε, όλα τα, όλους τους στόχους της πολιτικής για το φύλο. Επίσης, θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε το πρόγραμμα Δάφνη και όλα τα προγράμματα που θέλουν να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών και δεχόμαστε τις κριτικές που ασκήθηκαν πως είχαμε μια βασική μείωση των κονδυλίων που είναι διαθέσιμα για το Δάφνη τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύουμε πως όλα τα ταμεία που έχουν να κάνουν για την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών θα πρέπει να αξιολογηθούν έτσι ώστε να λάβουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι πετυχαίνουμε κάθε φορά. Εμείς δεν συμφωνούμε με κάποια από τα θέματα που έθιξε η έκθεση. Καταρχήν, η παραπομπή στην κρίση του 2008 που μιλάει για υποχώρηση σε σχέση με την ισότητα, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί με έναν τρόπο να είναι ισορροπημένος και μη ιδεολογικός. Δεύτερον, η πληθώρα των ευρωπαϊκών ε, οργάνων που ασχολούνται με θέματα γυναικείων δικαιωμάτων και άλλα συναφή. Νομίζω ότι το Ινστιτούτο που έχουμε είναι αρκετό και θα πρέπει να το στηρίξουμε και να το βοηθήσουμε και όχι να δημιουργήσουμε και να πολλαπλασιάζουμε τα σχετικά όργανα. Δεν θεωρούμε πως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμόδιο για να χρηματοδοτεί ε, αυτά τα Ινστιτούτα σε επίπεδο κράτους μέλους και δεν θέλουμε η αρχή της ισότητας να οδηγήσει σε διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις ε, που συμμετέχουν σε project τα οποία εν μέρη χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίσης, θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα της ε, προϋπολογιστικής διαδικασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνεται υπόψη το φύλλο, αλλά ε, σύμφωνα με κάποιους στόχους που θα αξιολογούνται, δηλαδή όπου υπάρχει αντικειμενική ανάγκη για παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ταμείων της ήδη περνά από ένα είδος pre-screening έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε πως δεν υπάρχουν διακρίσεις που να εξαρτώνται από το φύλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις ή αμφιβολίες σας παρακαλώ πολύ να τις απευθύνετε στην Μπάρμπαρα Ματερά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βυσνιέσκα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ασχολείται με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει να αντιμετωπίσει ποτέ είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτήν και δυστυχώς η έκθεση την οποία προετοίμασε η συγγήτρια δεν πρόκειται να βελτιώσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πολιτών, γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι πιο διάφανος και πιο αποτελεσματικός. Είναι δύο στοιχεία αυτά τα οποία λείπουν από τα ευρωπαϊκά α, ταμεία. Και όταν μιλάμε για ισότητα μεταξύ φύλων, να σας πω πως τα τελευταία χρόνια ο προϋπολογισμός για τα θέματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως ένα πολύ ακριβό εργαλείο για να προωθηθούν τα φεμινιστικά ε, ζητήματα και νομίζω πως ε, θα πρέπει να τα σκεφτούμε τα θέματα αυτά, αλλά να λάβουμε υπόψη πως ε, εδώ μεγάλες αλλαγές εμείς δεν μπορούμε να εισάγουμε. Και σήμερα το να βάλουμε το στοιχείο του φίλου σε όλες τις πολιτικές με έναν τρόπο που προκαλεί σύγχυση και που δεν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και ακριβής, το μόνο που θα κάνει είναι να ε, μειώσει ακόμα ε, τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα στα μάτια του πολίτη. Τώρα το να ψάχνουμε για την ισότητα έτσι δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει γιατί τέτοιου είδους λύσεις τελικά φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα και δεν νομίζω πως είναι η καλύτερη τακτική για να επιλέξουμε. Καλύτερα λοιπόν θα ήταν η ισότητα αυτή να βασίζεται στις ικανότητες που έχει κάθε άτομο, γιατί η ισότητα μεταξύ φίλων με τον τρόπο που το περιγράφεται θα οδηγήσει σε χρηματοδότηση όλων των ειδών ε, έργων, ενώ θα έπρεπε να χρηματοδοτούμε μόνο αυτά που θα κάνουν πραγματική διαφορά. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, θα πρέπει να στοχεύσουμε περισσότερο στην πάταξη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για το να ε, χτίσουμε ε, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία που θα επιτρέπουν στις γυναίκες να είναι απόλυτα ενταγμένες στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για την πρόταση, την κατάθεση της έκθεσης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτές τις επεξηγήσεις. Εμείς οι πράσινοι χαιρετίζουμε αυτό το σχέδιο και σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούμε. Είναι πολύ καλό αυτό το οποίο εκθέσατε. Ήδη στο πρώτο τμήμα της έκθεσης. Σαφώς και τα όσα αναφέρονται σε σχέση με την εφαρμογή ή την μη εφαρμογή σε σχέση με την ολοκλήρωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές και η κατεύθυνση είναι σαφής για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου. Ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα πρέπει να αναφερθούμε θετικά αναφερόμαστε στο gender budgeting, όπως ε, σε πολλά σημεία της έκθεσης αναφέρεται. Εδώ θα κάνουμε κάποιες συμπληρώσεις για το gender budgeting από πλευράς μας, με τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό, το gender budgeting, ένα μέσο κλειδί για την ισότητα των φύλων και την δίκαιη κατανομή κονδυλίων στα φύλλα. Εδώ και χρόνια ζητάμε το gender budgeting από τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μέχρι σήμερα όμως αδράνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο gender budgeting σε όλα τα κονδύλια. Και όπως σήμερα είπατε θα πρέπει να αλλάξει αυτό και όχι μόνο για εκείνα τα προγράμματα που είναι πιο προφανές αυτό. Είναι αυτονόητο ότι υποστηρίζουμε την εισηγήτρια για την εφαρμογή συγκεκριμένων δικτών όσον αφορά τα φύλλα και monitoring και αξιολόγηση όλων των μέτρων στη συνέχεια που αφορούν μέτρα που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του προϋπολογισμού. Και επεκτείνουμε αυτή τη διεκδίκηση, αυτή την απέτηση για μια εξ άντε αξιολόγηση, εκ προημίου, εκ των προτέρων αξιολόγηση. Σε, επίσης στον τομέα της παρουσίασης ε, των, ε, της σπουδαιότητας ε, των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την γενική ισχύ αυτών των μέτρων από πλευρά κονδυλίων σύμφωνα με δείκτες ανάλογα με το φύλλο που είναι απόλυτα αναγκαίοι και για την χρήση του Ταμείου περιφερική Ανάπτυξης να δούμε τι γίνεται ιδιαίτερα για τη σπουδαιότητα κοινωνικών υποδομών για την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη για θεσμούς και φορείς για τη μέρημνα των παιδιών και τον ορίζοντα 2020 και το νέο στρατηγικό ταμείο επενδύσεων Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την πολιτική επενδύσεων ή τη νέα κατεύθυνση της πολιτικής επενδύσεων και τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστούμε για την έκθεση. Προσβλέπουμε στην ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Χανιμπόλ έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Κλέα για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ καλό το ότι έχουμε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή μια τόσο σαφή και άμεση κατεύθυνση να θέτουμε τον προϋπολογισμό gender budgeting στο επίκεντρο με αυτή την κατεύθυνση. Κάναμε λόγο και κάνουμε λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα για αυτά και τώρα υπάρχει ένας τρόπος να αρχίσουν να λειτουργούν όλα αυτά. Και είναι πολύ καλό το ότι η Κλέρ εξέτασε τα τρία προγράμματα και τα υπογράμμισε στην ε, σπουδαιότητα και εμβέλειά τους. Και ήταν σε θέση να πει ότι θα έπρεπε να είμαστε σε θέση σε αυτά τα προγράμματα να εντάξουμε το gender budgeting. Φυσικά όταν συντάσσει κανείς μια τέτοια έκθεση, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαιτείται και από πλευρά συζητού τα κυριότερα σημεία επιλέγονται στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Πολλά μας ενδιαφέρουν και τα ακολουθήσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα θέλω να προτείνω εδώ ότι θα έπρεπε επίσης ε, να εντάξουμε κάτι για τους πρόσφυγες σε αυτό το πλαίσιο και μπορούμε να το κάνουμε με μια τροπολογία για παράδειγμα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αναφορά για ένα ταμείο για τα φύλλα ή διάθεση κονδυλίων ανάλογα με το φύλλο για πρόσφυγες. Όπως γνωρίζουν τα μέλη, ήμουν πρόσφατα εισηγήτρια για αυτό το θέμα σε μια έκθεση. Και είναι σαφές ότι υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να κάνουμε επιτακτικά ό,τι περνά από το χέρι μας για τους πρόσφυγες, γυναίκες και παιδιά που είναι μόνες τους και μόνα τους και όταν έρθει η χρονική στιγμή που μπορούμε να το κάνουμε, να καταθέσουμε μια τροπολογία για να ενδυναμώσουμε αυτό το πλαίσιο. Το χρειαζόμαστε αυτό για να γίνει ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κυρία Χάνιμπορ. Δεν ξέρω, θέλει η κυρία να απαντήσει στις παρεμβάσεις που έγιναν σε σχέση με την έκθεση. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σας. Πολλά από αυτά πιστεύω ότι φυσικά θα πρέπει να τα εκπονήσουμε και να τα επεξεργαστούμε στις συναντήσεις και οδών εισηγητών. Υπάρχει σαφώς αυτή η πρόπτικη για το νέο έτος. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που συμφωνούν με την εκθεσή μου φυσικά. Αυτονόητο είναι. Δίνοντας συνέχεια σε κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν, για παράδειγμα σε σχέση με την κρίση του 2008 και τις επιπτώσεις που είχε αυτή η χρηματοοικονομική κρίση στις γυναίκες. Αναπόφευκτα δεν συμφωνώ σε σχέση με το ότι δεν υπήρξε λέει σε σχέση με κάποια μελέτη, κάποια επίπτωση. Υπήρξαν μελέτες σχετικά και υπάρχουν επιπτώσεις και πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτά στις συναντήσεις και οδών εισηγητών. Και κάτι άλλο Κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα του να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά σε σχέση με τους πολίτες ε, στο πρώτο κατώτατο επίπεδο μεταξύ των πολιτών. Πολλά μπορούν να γίνουν για να υποστηριχθεί αυτό που βρίσκεται υπό εξέλιξη μεταξύ των πολιτών και κάποια από αυτά τα σημεία θα τα συζητήσουμε και θα τα διαβουλευτούμε επ' αυτόν με τους σκιώδεις εισηγητές στο μέλλον. Ουσιαστικά δεν εκπλήσει κανένα ότι για τα θέματα που ε, πρέπει να εξεταστούν ε, αφήνουμε μερικά θέματα για να τα δούμε ξεχωριστά. Και προφανώς ε, προσβλέπω στο να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, το σημείο εξάντα για την αξιολόγηση που αναφέρθηκε και ιδιαίτερα όπως είπε η Μέρη υποστήριξη των προσφύγων, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μόντι. Τώρα για να σας πληροφορήσω προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 9 Δεκεμβρίου θα λήξει 12 το μεσημέρι. 9 Ιανουαρίου 2017 θα εξεταστούν οι τροπολογίες. 25 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε την έκθεση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και προβλέπεται για τον Μάρτιο 2017 να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004 ε, σε σχέση 2144 ε, για την ισότητα των φύλων κονδυλίων, από πλευρά κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχετε τον λόγο συνάδελφε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες, Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την ανάπτυξη των τελευταίων στοιχείων έχουν κατατεθεί πάρα πολλές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για όλες. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμες νομίζω ότι συνεισφέρουν στην ποιότητα της έκθεσης. Να ευχαριστήσω επίσης τους Κιώδης και όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Με αφορμή αυτό να πω ότι βασικός στόχος της έκθεσης είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας και της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των τομέα παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει εμείς να αποδυναμώσουμε ε, την, ε, ε, τον στόχο αυτό. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες έχουν σαν κεντρικό στόχο την διεύρυνση των πεδίων τα οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί. Δηλαδή χρηματοπιστωτικός τομέας, πρόσβαση στις βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο είναι βασικό για την επιχειρηματικότητα των γυναικών και αντιμετώπιση των στερεοτύπων για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Έχουμε μία συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με τον τομέα των ασφαλιών και οι τροπολογίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Κάποιες ξεπερνούν βέβαια την εμβέλεια της έκθεσής μου πολλές τροπολογίες αφορούν την αγορά στην αγορά εργασίας. Εδώ υπάρχουν άλλες οδηγίες οι οποίες ρυθμίζουν το θέμα της ισότητας των φύλων. Γι' αυτό ακριβώς και οι τροπολογίες αυτές δεν θα έπρεπε να μας αφορούν. Υπάρχουν οδηγίες επίσης για την αναθεώρηση και τη διεύρυνση του στόχου της ε, ε, οδηγίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαφήμιση σαν παράδειγμα η τόσο σημαντική για την οικονομία είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών. Άμεσα λοιπόν νιώθει κανείς την ανάγκη να εφαρμόσει ε, τις οδηγίες αυτές και σε άλλους τομείς. Από την άλλη βέβαια τα μέσα αυτά υπόκεινται στην αρχή της επικουρικότητας ως εκ τούτου δεν είμαι βέβαιος αν μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε εδώ. Πάντως η απλή σύνδεση ανάμεσα στην διαφήμιση και τις υπηρεσίες είναι σαφής και αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε στις επόμενες ε, συναντήσεις μας. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες για την εφαρμογή της λεγόμενης οριζοντίας οδηγίας και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη οδηγία έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης πολυετούς και οι περισσότερες χώρες είναι κατά. Και αυτό όμως θα το συζητήσουμε. Και τέλος υπάρχουν τροπολογίες ε, σχετικά με την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εγώ είμαι κατά των τροπολογιών αυτών, αν και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι κείμενο θα έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρ' όλα αυτά θεωρείται ότι είναι το επίπεδο αναφοράς της καταπολέμησης της βίας. Θέλουμε λοιπόν να αποκτήσει σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι συζητιέται η συγκεκριμένη πρόταση και πιστεύω ότι εν πάση περιπτώσει τα τμήματα της οδηγίας που άπτονται της ασφάλειας των γυναικών στον τομέα των μεταφορών σαν παράδειγμα είναι ο σωστός τομέας για να αναφέρουμε ε, την συγκεκριμένη σύμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρέγνα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Εισηγήτρια και αγαπητές σκιώδεις εισηγήτριες. Θα ήθελα κάποια πράγματα να πω σε σχέση με αυτές τις παρατηρήσεις και να προσθέσω ή να απαντήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση μου αρέσει προσωπικά πολύ. Πολλές σημαντικές πτυχές ε, καλύπτονται. Ωστόσο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συχνά απουσιάζουν τα συμπεράσματα όλων αυτών των θέσεων. Τώρα, ως Ευρωβουλευτές θα έπρεπε έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών συγκεκριμένες εντολές ή τέλος πάντων κατευθύνσεις να εκπονήσουμε και να τους δώσουμε. Και οι συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα συμπεράσματα εδώ προς τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή απουσιάζουν πολλαπλά στην έκθεση και θέλω αυτό να αποσαφινιστεί και να καλυφθεί. Αναφέρθηκε η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, Ιστάνμπουλ για το θέμα δηλαδή της διεκδίκησης της ε, απέτησης να κυρωθεί, να επικυρωθεί. Δεν βρίσκω όμως το λογικό συμπέρασμα. Δηλαδή, σε σχέση με αυτή τη σύμβαση αναφέρεται μεν, αλλά θα έλεγα ότι μια σημαντική σύμβαση όπως η της Κωνσταντινούπολης όχι μόνο πρέπει να τονίζεται η σπουδαιότητά της, αλλά αντίστοιχα θα πρέπει να δίνεται η εντολή δράσης ώστε να καλυφθεί η ανάγκη να ακυρωθεί και να προαχθεί. Άλλο θέμα σε σχέση με τα δίκαια και τις εφαρμογές των κρατών μελών. Υπάρχουν διαφορές και είναι ανησυχητικό αυτό όταν βλέπουμε ότι η προσπάθεια, η προστασία έναντι ε, αρνητικής ε, διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να δημιουργήσει υψηλής προδιαγραφής ε, συνθήκες, όρους και προϋποθέσεις για την προστασία αυτή. Οι υπηρεσίες για την ισότητα των φύλων έχουν διαφορετικό εξοπλισμό και κονδύλια στα κράτη και δεν μπορούν παντού να είναι ανεξάρτητες όπως θα έπρεπε. Το, αντίστοιχες τροπολογίες προέρχονται και από, άλλα, από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Είδα μερικές ε, από μια συνάδελφο. Ελπίζω ότι η ενίσχυση της ε, ισότητας ε, των γυναικών θα επιτευχθεί. Πρέπει να είναι αποτελεσματική αυτή η φορείς και ανεξάρτητη στη δράση τους και πρέπει να έχουν και αρκετά κονδύλια με τα οποία θα πρικιστούν για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ψηφιοποίηση. Είναι και αυτό ένα σημείο που πρέπει να αναφερθεί. Σε σχέση με το 2004 βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον σήμερα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για την ισότητα και τις υπηρεσίες και την, και την δράση που όχι μόνο αναλογικά αλλά ε, και ψηφιοποιημένα θα πρέπει να δράσουμε. Ας είμαστε πιο ε, συγκεκριμένοι για τα θέματα ευθύνης για παράδειγμα που πρέπει να καλύπτεται. Εδώ και η νομική επιτροπή δραστηριοποιήθηκε σχετικά. Είναι σημαντικό το αίτημα να καλυφθεί και αυτή η πτυχή. Τέλος διαφήμιση. Διαφήμιση στα μέσα όσον αφορά και την προετοιμασία προετοιμασία, κατάρτιση. Γνωρίζω ότι πολλαπλά έχει συζητηθεί το θέμα αυτό και ε, αφαιρέθηκε, εξαιρέθηκε ρητά από την οδηγία. Πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη θλίψη τους γι' αυτό και υπάρχουν τροπολογίες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ήδη κατά το παρελθόν το 2004 είχαμε δει ότι ήδη τότε δημιουργούσε ένα μείζον πρόβλημα αυτή η κατάσταση σε σχέση με τη διατύπωση και την μη συμπερίληψη κάποιων πραγμάτων. Να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, πραγματιστές, αλλά εκεί όπου πρόκειται για κλασικούς ρόλους για τα φύλλα ή τα πρόσωπα, θα πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές δυνατότητες για τα κλασικά συμβολικά ε, δρόμενα των ρόλων. Θα πρέπει να είμαστε πιο διαφοροποιημένοι. Και τέλος, ε, για τα επαρκή στοιχεία που πρέπει να διασφαλίζονται. Θα πρέπει εδώ στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητηθεί να είναι πιο αποτελεσματικά και πιο αποτελεσματικοί. Να παρέχονται στοιχεία για τη σωστή αξιολόγηση, δηλαδή σε σχέση με την ε, αρνητική μεταχείριση πρέπει πολλαπλά να αντιμετωπιστεί. Έχουμε τροπολογίες λοιπόν για να συμπληρώσουμε αυτά που αναφέρθηκαν πιο πριν. Και ευελπιστώ ότι η μία ή η άλλη θα κατατεθεί έτσι και θα εγκριθεί. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει ζητήσει τον λόγο να παρέμβει. Έτσι λοιπόν, αν η κυρία Κολόσκα θα ήθελε να απαντήσει σε αυτές τις παρεμβάσεις, σε κάποιες ερωτήσεις. Η ολοκληρώνουμε τη συζήτηση όπως επιθυμείτε κυρία. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Ε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια της προσπάθειας πλήρους εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι η ανεπαρκής, θα έλεγα, εφαρμογή. Μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία μια οδηγία, αλλά στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Αυτό λοιπόν είναι βασικό πρόβλημα. Η ανταλλαγή λοιπόν χρηστών πρακτικών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί σαν στόχος. Και η παρακολούθηση και οι παρατηρήσεις γύρω από αυτό το θέμα από πλευράς των κρατών μελών είναι καλοδεχούμενες. Αλλά ακόμα και αν ε, δεν έχει επικυρωθεί από όλες τις χώρες, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της βίας. και θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επίπεδο στο οποίο θα εφαρμοστούν οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων. Η έκθεση λοιπόν περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά θέματα. έτσι ώστε να υπάρξει κατάλογος όλων των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων γύρω από τις διακρίσεις στις χώρες μέλη. Η ψηφιακή πραγματικότητα περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή αλλά με ανεπαρκή τρόπο και γι' αυτό εμείς θα βάλουμε άλλα δύο σημεία Πρώτον, η ψηφιοποίηση της αγοράς έχει οδηγήσει ανάμεσα σε άλλα και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών τομέων. Η καταμεριστική οικονομία, όπως επίσης και ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Airbnb για την ενοικίαση κατοικίας, καταλήμματος, είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον. Θα έχουμε πολύ περισσότερα τέτοια παραδείγματα στο μέλλον. Ως εκ τούτου λοιπόν τίθεται το θέμα της ασφάλειας των γυναικών όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Για τις, για τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο διαδίκτυο Βλέπουμε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμα περισσότερο από τις άνδρες και εδώ χρειάζεται να υπάρξει ε, μια επιμέρους προσπάθεια. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να εργαστούμε σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να συλλέγονται και να ταξινομούνται με κριτήρια φύλου και να υπάρξει εφαρμογή της ίδιας ακριβώς μεθοδολογίας για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε ακριβώς τα δεδομένα και δεν θα καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα. Πάντως το θέμα της διαφήμισης πρέπει να τεθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κοντλόφσκα. Εδώ τελειώνει το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο. Προσβασιμότητα σε ε, προϊόντα και υπηρεσίες. Η κυρία Λεγκρίπ θα εκπροσωπήσει την εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά καλούμε την τελευταία στιγμή να αντικαταστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Φαραγκούτ, η οποία έπρεπε να λείψει, δεν είχε προβλεφθεί όμως η απουσία της. Έχουν προετοιμαστεί λοιπόν κάποια τμήματα προτάσεων τα οποία θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας όχι τη μητρική γλώσσα, ούτε και τη γλώσσα της κυρίας Φαρακούτ, αλλά θα σας τα διαβάσω ή στην αγγλική γλώσσα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν από κοινού να δούμε το πώς έχουν ε, στην παρούσα φάση οι συνθήκες και να δούμε ποιες είναι οι τροπολογίες οι οποίες έχουν προταθεί και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων για τις 151 τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο είχε ε, προετοιμάσει η κυρία Φαραγκούτ 19 τροπολογίες ε, ΕΛΚ, 21 σοσιαλιστών 4 φιλελευθέρων, 26 των συντηρητικών, 59 τροπολογίες της Γκουε, 4 τροπολογίες των Πρασίνων και 14 τροπολογίες των μη εγγεγραμμένων. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα πρέπει κανονικά να γίνει στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τι μπορεί κανείς να πει στην παρούσα φάση για τις διάφορες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί ήδη. Καταρχάς, απαιτήσει προσβασιμότητας. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι οι απαιτήσει αυτές συναδεύονται στο παράρτημα με ακόμα πιο υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας. Πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των προσώπων με αναπηρία και γυναικών με αναπηρία ε, και ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Ε, Απαιτήσει σε επίπεδο ε, εγκαταστάσεων όπου δεν είναι επαρκής για την χρήση από πλευράς της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών το, οίκη, το <clears throat> κτιστό περιβάλλον θα λέγαμε, το δομημένο περιβάλλον πολλές φορές δεν καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι προσβάσιμες ε, οι εγκαταστάσεις αυτές. Τώρα, για τις ε, σημασία που έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία αυτή. Information on the accessibility characteristics of the products Ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια και όχι εφόσον έχουμε λάβει έτοιμα από την αρμόδια Εθνική Αρχή. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο σημαντικό για μας. Τώρα για το θέμα της παρακολούθησης της αγοράς, το άρθρο 17 δηλαδή, η ενημέρωση για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσει προσβασιμότητας θα πρέπει να δημοσιεύονται συστηματικά και όχι μόνο κατόπιν ετήματος. Για το θέμα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης, που είναι το άρθρο 25, Νομίζω ότι είναι θετικό και στο σχέδιο πρότασης για την οδηγία λέμε πως οι καταναλωτές είναι αρμόδιοι, όπως επίσης και οι διάφορες οντότητες, οι ενώσεις καταναλωτών ή και δημόσιοι φορείς που μπορούν να καταγγείλουν αυτές τις υποθέσεις σε αρμόδιους φορείς. Όμως, επειδή πολλές φορές τα άτομα αυτά έχουν δυσκολία πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δεν είναι αρκετό αυτός διάταξη για να κατλήψει όλες τις περιπτώσεις που θέλουμε να προσφύγουμε κατά του κατασκευαστή. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει ε, να εστιάζουμε στην αγωγή του καταναλωτή και τη συγκεκριμένη δράση του καταναλωτή, αλλά σε ένα ευρύτερο σύστημα ε, που θα καλύπτει και αυτές τις διαστάσεις. Θα πρέπει δηλαδή να έχει δυνατότητα η συγκεκριμένη υποπτεύουσα αρχή να ε, παρακολουθεί και την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας. Τώρα, άρθρα 26 ε, κυρώσεις τα τέλη τα οποία συλλέγονται θα πρέπει να επενδύονται σε μέτρα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πληρωμή των κυρώσεων να θεωρείται ως μια φθηνή εναλλακτική για να μην εφαρμόζονται οι απαιτήσει που περιγράφονται στο άρθρο 3. Ελπίζω πως αυτές οι γενικές ανησυχίες και τα σχόλια αυτά για όλα τα θέματα που προκύπτουν να είναι επαρκή. Με συγχωρείτε που σε κάποια στοιχεία δεν ήμουν απόλυτα σαφής, αλλά θα καταλάβατε φαντάζομαι πως ε, επειδή πήρα τη σκητάλη μάλλον τελευταία στιγμή από κάποια συνάδελφο, δεν ήμουν σε θέση να εμβαθύνω πάρα πολύ σε κάποια από αυτά τα θέματα και θα ήθελα να ε, σας ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η, η κυρία Φαραγκούτ ήθελε να, ε, θα ήθελε να επαναλάβω πως σας ζητά συγγνώμη για αυτό που συνέβη, αλλά είναι ξεκάθαρο και η συγγήτρια μας είχε καιρό να το πει, είχε, είχε πολλές φορές την ευκαιρία να το πει αυτό. Ε, εμείς ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στεκόμαστε στο θέμα και παρακολουθούμε ε, με ιδιαίτερη φροντίδα αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να τη βελτιώσουμε και να είναι ακόμα πιο λειτουργική και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των συμπολιτών μας που έχουν δυσκολίες πρόσβασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση με τις ε, διάφορες πολιτικές ομάδες. Κυρία Χέτη, παρακαλώ, πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχήν την εισηγήτρια που δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραστεί Ευχαριστώ για αυτό το σχέδιο. Ήταν ενδιαφέρον και όλες οι τροπολογίες ήταν ενδιαφέρουσες, οι τροπολογίες που κατατέθηκαν. Σε αυτή τη χρονική στιγμή μια σημαντική, μια αποτελεσματική γνωμοδότηση πρέπει να δημιουργηθεί και σε σχέση με τη γνωμοδότησή μας πρέπει να αναφέρονται οι πτυχές της ισότητας με κάθε τρόπο και να επισημαίνεται ότι υπάρχει πολλαπλή αρνητική διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τις γυναίκες με ειδικέ ανάγκες. Η πτυχή της ισότητας πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη. Ποτέ δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η ενιαία εσωτερική αγορά αν δεν συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ε, κοινωνικά σε αυτήν. Και αυτό απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα από εμάς. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να αγνοούμε τα προσκόμματα και τα εμπόδια. Πρέπει να απαιτήσουμε την ισότητα, να επιτευχθεί η ισότητα. Πολλές τροπολογίες στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθούν δηλαδή προϋποθέσεις ώστε μια πλήρη συμμετοχή στην ενιαία εσωτερική αγορά να επιτευχθεί για όλους τους πολίτες. Και αυτό να αντιμετωπίζει και την πολλαπλή αρνητική διακριτική μεταχείριση που αφορά άτομα με μειονεξίες, άτομα με ειδικέ ανάγκες και σε σχέση με το πλαίσιο της εντολής της ε, Κοινοβουλικής μας Επιτροπής πρέπει να το τηρήσουμε. Κάποιες από τις τροπολογίες προφανώς είναι καλές σε σχέση με τη διαπίστωση, διατύπωσή τους όμως δεν εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων αυτό που ανέφερα της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη ώστε η γνωμοδότησή μας να είναι αποτελεσματική και ισχυρή, να μπορέσει να ασκήσει επιρροή. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία με την εισηγήτρια και τις άλλες σχεώδεις εισηγήτριες και θα έλεγα ότι πραγματικά έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε τον, τη μάχη για την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ.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 Dobre, takže ešte raz, už máte preklad? Ακούτε, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Je preklad zo Slovenčiny zabezpečený? Υπάρχει διερμηνία από τα Σλοβακικά. C'est bon Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι να το ξαναπροσπαθήσουμε. Ο αριθμός των τροπολογιών 150 μία τροπολογίες και το περιεχόμενο των τροπολογιών αυτών καταδεικνύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί αυτή η πρόταση να έχει ένα φιλόδοξο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί. Κάποιες ε, προτάσεις ε, τροπολογίας θέλουμε να διατυπώσουμε ώστε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές για παράδειγμα ή αυτόματες συσκευές, αυτόματα να μπορέσουν να ενταχθούν όμως υπάρχουν και περιορισμοί από πλευράς ε, θεμάτων ουσίας και όπως αναφέρθηκε καλό θα ήταν ε, φιλοσοφικά να μπορούσαμε να πετυχαίναμε μια αλλαγή της κατεύθυνσης. Η οδηγία αυτή δεν πρέπει να αφορά μόνο άτομα με ειδικέ ανάγκες, πρέπει να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες και όχι μόνο εκείνους που έχουν κάποια μειονεξία. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία θα συνεισφέρει στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και εδώ δεν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο νομοθετικά αυτούς τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος τρόπος ε, ένταξής τους, να έχουμε μια ολοκληρωμένη κοινωνία που θα συμπεριλαμβάνει σφαιρικά όλους τους πολίτες και έτσι, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε τις τοπολογίες. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κούνεβα έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις προηγούμενες εισηγητές. ο μερικά σύντομα σχόλια από την πλευρά μου. Η οδηγία δεν έχει συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου Στι προτάσει για την προσβασιμότητα στι υπηρεσίε και τα προϊόντα. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Γιατί υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια γυναίκε και κορίτσια με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτέ σύμφωνα με τα στατιστικά κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε συνθήκε φτώχεια. Επίση έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε τέσσερι εργασία, στην εκπαίδευση, σε πολιτιστικά γεγονότα και άλλα. Και όπω διαπιστώνει στην γνωμοδότηση τη η σάδελφο Φαραγκούτ, δεν είναι επαρκής οι απαιτήσει για το δεδομένο περιβάλλον. Όμω, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα το δεδομένο περιβάλλον. εκτό από προϊόντα και υπηρεσίε Προσβάσιμε σε γυναίκε και κορίτσια. Να σα πω ένα παράδειγμα. όσε έχουν υποστεί βία μπορούν να καλούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό για να αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη. Τι γίνεται όμω με τι γυναίκε που έχουν αναπηρία που επηρεάζουν την ομιλία του, πώ μπορούν αυτέ να αναζητήσουν άμεσα βοήθεια. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να μοιραστώ έρχεται από το χώρο της εργασίας. Σε πολλά από τα κράτη-μέλη γίνονται προσλήψεις ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες κρατικές υπηρεσίες. Όμως, συχνά τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες δεν είναι φιλικές για χρήση από άτομα με αναπηρία. Αποκλείουμε δηλαδή μέσα στο ίδιο το περιβάλλον τις εργασίας που ένα άτομο με αναπηρία. Μερικές από τις προτάσεις για να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία είναι οι εξή. Πρώτο, το δεδομένο περιβάλλον να είναι φιλικό και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Δεύτερον, τα ευρέως χρησιμοποιημένα προϊόντα όπως για παράδειγμα τα ρολόγια, τα μαξίδια, τα κρεβάτια, εξετάσεις των γυναικολόγων, τα προϊόντα αντισύλληψης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άτομα με αναπηρίες. Τρίτον, οι υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής υγιεινής υποστήριξης μητερών και παιδιών θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες από όλες και όλους. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις σκέψεις μου Τις υπόλοιπες τις έχετε δει και μέσα από τις τροπολογίες. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια και τους συνάδελφους. Φαντάζομαι θα καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές τροπολογίες που θα αναδεικνύουν την διάσταση του φύλου στην οδηγία και την προσβασιμότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, eh, Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούνεβα. Δεν ξέρω η κυρία Λεγκρίπ θέλει να αναφερθεί, να απαντήσει κάτι. Όχι. Ωραία. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η χορήγηση απαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2015 για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και του Ιδρύματος για την ισότητα των φύλων. Αν συμφωνείτε θα διεξαχθεί η κοινή συζήτηση επ' αυτών όπως και σε άλλες, με άλλες αφορμές από πλευράς εισηγητού η εισηγήτρια είναι η κυρία Νταντσίλα που δεν παρίσταται και από πλευρά τη ε, συναδέλφου θα την αντικαταστήσει συνάδελφο στην παρουσίαση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την κυρία Νταντσίλα που έχει συντάξει την γνωμοδότηση για τον Γενικό προπολογισμό της Ένωσης και της Επιτροπής και έπρεπε να παρουσιάσει αυτή την παρουσίασή της, δεν μπορεί όμως να παραστεί για την χορήγηση απαλλαγή για το συνολικό σχέδιο του προϋπολογισμού τονίζει η εισηγήτρια ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικών και στο gender budgeting και σε όλες τις φάσεις του προϋπολογισμού και στο μεσοπρόθεσμο χρηματοοικονομικό πρόγραμμα πρέπει να εντάσσεται. Η γνωμοδότηση τονίζει ότι μετρήσιμοι δείκτες πρέπει να υφίστανται για τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα των μέτρων του σχεδίου προϋπολογισμού για την ισότητα στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση του προϋπολογισμού. Δείκτες που θα συνάδουν με τη στοχοθέτηση και την, τα, κέντρα, τα κέντρα βάρους ε, των προσπαθειών. Παρόλη αυτή την τοποθέτηση για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να έχουν ληφθεί. Γι' αυτό ζητούμε να υπάρξει μια αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης όλων αυτών στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Ζητεί επίσης η γνωμοδότηση από το ελεγκτικό συνέδριο στο, ε- στην ετήσια έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο να αναφέρεται σε συγκεκριμένα θέματα φύλου που αφορούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει δηλαδή εδώ κάτι το οποίο επανειλημμένα και πολλαπλά θα εξετάζεται. Ιδιαίτερα για τα δίκαια και την ισότητα των πολιτών της Ένωσης που θα συμπεριλαμβάνει και τους στόχους του προγράμματος Δάφνη οι στόχοι επαναλαμβάνονται όσον αφορά τη στοχοθέτηση που το πρόγραμμα για την ηθαγένεια και την ισότητα RWC ε, ε, και την ισότητα καθώς επίσης και την δίκαια κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των διαφορετικών τομέων που εντάσσονται στους συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος. Διότι στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας σε σχέση με τους στόχους της Δάφνης, του προγράμματος Δάφνης, λιγότερα κονδύλια δόθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα 2007-2013. Η συντάκτη της γνωμοδότησης εδώ εκ νέου τοποθετείται με σαφήνεια ότι χρειάζονται ξεχωριστά κονδύλια για την ισότητα των γυναικών και σε σχέση με το 13881 κάθετος 13 για το πρόγραμμα για την ηθαγένεια και την ισότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια να υποβάλει μια έκθεση παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 14 εδάφιο 2 <clears throat> και με τους δείκτες, μετρήσιμους δείκτες για την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μέτρων. Δηλαδή μια ετήσια έκθεση που ετήσια θα συντάσσεται για να μπορεί να παρακολουθεί κανείς την εποπτεία όλων αυτών. Για την εκπόνηση της γνωμοδότησης <clears throat> αυτή την έκθεση εποπτείας για το 2015 δεν μπορέσαμε να την αποκτήσουμε. Δεν δόθηκε αυτή. Ζητείτε εδώ λοιπόν να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να μας διατεθεί αυτή η έκθεση τα μέλη ευρωβουλευτές προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και να καταθέσουν τροπολογίες. Προθεσμία καταληκτική για τις τροπολογίες είναι 6 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Η κυρία Λεγκρίπ θέλει να παρέμβει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ήθελα καταρχήν να εκφραστώ εκ μέρους της Μπάρμπερα Ματερά για να μιλήσει για το θέμα της απαλλαγής ε, εκ μέρους του ΕΛΚ. Είναι σε άδεια μητρότητας αυτή τη στιγμή, οπότε έχει πραγματική δικαιολογία για το γεγονός και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή που δεν είναι κοντά μας και μου ζήτησε να πω δύο λόγια τα οποία θα πω στα αγγλικά και πάλι. Εγώ είμαι σαφέστατα υπέρ της χρήσης των γαλλικών και της γαλλοφωνίας, αλλά χρειάζεται για το λόγο αυτό, επειδή μεταφέρω τα λεγόμενα της κυρίας Ματερά, να μιλήσω στα αγγλικά. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια για την πολύ συγκεκριμένη αυτή ε, γνωμοδότηση και το, την καλή της δουλειά που έκανε σχετικά. Η κυρία Ματέρα χρόνια ασχολήθηκε στην Επιτροπή μας, όπως επίσης και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για το θέμα αυτό και κυρίως ασχολήθηκε με το θέμα των, της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών και για να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και για να βοηθήσουμε για τα όσα έχουν ήδη προταθεί, νομίζω πως θα πρέπει να εστιάσουμε στους συγκεκριμένους στόχους και όχι να ζητάμε η ισότητα των φύλων να λαμβάνεται υπόψη με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις πολιτικές. Γιατί Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί διαφορετικά αν προσπαθούμε να το εντάξουμε εγκάρσια σε όλες τις πολιτικές, τότε ίσως να μην φανούμε ρεαλιστές και ενδεχομένως να κατηγορηθούμε πως κυνηγάμε ουτοπίες. Εμείς ως ΕΛΚ θα πρέπει να προτιμήσουμε να μην συμπεριλαμβάνουμε σε όλες τις πολιτικές ε, τη διάσταση της ισότητας των φύλων, αλλά να ζητήσουμε σε κάθε περίπτωση να γίνεται μια αξιολόγηση μια αξιολόγηση των επιπτώσεων σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή να στοχεύουμε καλύτερα και να βλέπουμε την επιπτωσιολογική μελέτη σε πιο πολύ βάθος. Και για να το πετύχουμε αυτό ε, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να αξιολογήσουμε το gender budgeting σε, οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε χώρο προκύπτει αυτό. Για να κλείσουμε και οποιασδήποτε ε, και οποιαδήποτε κενά έχουν ε, παραμείνει. Σας ευχαριστώ πολύ και αυτό θα προσπαθήσει να πετύχει και η κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βάνε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια κυρία Ντανσίλα για τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης και την εξαιρετικά καλή συνεργασία. Σε όλα τα σημεία συμφωνούμε ως πράσινοι. Σε όλα τα σημεία. Μόνο κάποιες συμπληρώσεις και ε, υπογραμμίσεις θα κάνουμε σε κάποια σημεία προς μια άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ενίσχυση του προϋπορισμού gender budgeting. Θα έλεγα όμως ε, η επικέντρωση της νομοδότησης θα πρέπει να είναι πιο έντονα εστιασμένη σε αυτό το gender budgeting. Διότι είναι πολύ δύσκολο διαφορετικά να αξιολογήσει κανείς αν τα κονδύλια συνεισφέρουν υπέρ της ισότητας ή όχι. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το gender budgeting και έτσι τα προσκόμματα και τα εμπόδια δεν μπορούν να, να ξεπεραστούν χωρίς ε, μια πιο ενισχυμένη εστίαση σε αυτά τα θέματα. Σημαντική είναι και η απέτηση να υπάρχει gender mainstreaming και η αναθεώρηση στο ενδιάμεσο διάστημα εμπεριέχεται μένα αλλά μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς και πιο κάθετοι. Επίσης στο σημείο 4 όπου οι στόχοι για το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 ορίζοντας 2020 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ή επιδόσεις. Πολλές φορές όμως κάποιοι είναι τυφλοί σε σχέση με την ισότητα και τους στόχους του 2020. Γι' αυτό θα πρέπει να διευρυνθούν καλύτερα και στα αγγλικά που ίσως είναι πιο εύληπτη η διατύπωση economy, effectiveness και efficiency, τα τρία ε ως άξονες. Εμείς οι πράσινοι λέμε αυτοί οι στόχοι πρέπει να διευρυνθούν κάπως ή να τροποποιηθούν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα, equality equity και ecology, τρία άλλα ε με διαφορετική κατεύθυνση, για να είμαστε υπέρμαχοι των στόχων αυτών, αλλά διαφοροποιημένα. Να υπάρξει δηλαδή μια διαφοροποίηση και διεύρυνση των στόχων για να πετύχουμε τα ευκταία και τα επιθυμητά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αν συμφωνείτε, που είναι και το τελευταίο στην ημερήσια διάταξή μας που είναι εκείνο που αναφέρεται στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για διακόπτη πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη. Σε μια πρώτη στιγμή είπα θα γινόταν κοινή συζήτηση για όλα αυτά σε σχέση με την αναφορά των θεμάτων φύλου Κυρία Νόελ, έχετε τον λόγο για την έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγής για το Ίδρυμα για την Ισότητα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά. Παίρνω και πάλι τον λόγο για την κυρία Ντανσίλα. Είναι η συγγήτρια για τη γνωμοδότηση για τη χορήγηση απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Για αυτά που θα ήθελα να εκθέσω, τα όσα σχετίζονται με την χορήγηση απαλλαγή και το σχέδιο γνωμοδότησης καθορίζει ότι η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρει ότι η οικονομική κατάσταση κατά τα τέλη του 2015 εμφανίζεται ικανοποιητική και σε σχέση με όλους τους υλικούς τομείς βαίνει καλώς και ε, δείχνει χρηστή χρήση των κονδυλίων. Επίσης οι προσπάθειες όσον αφορά την μείωση των ε, ε, ποσών που πρέπει να μεταφέρονται από έτος σε έτος η γνωμοδότηση κτιμά επενεί την αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος Ζητεί όμως μια καλύτερη χρήση του φόρουμ, του βήματος των πραγματογνωμόνων, ώστε να υπάρχει, να συνάδει με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης η συντάκτρια γνωμοδότησης ε, αναφέρει επιπλέον ότι χαιρετίζουμε κατά τα άλλα την επέκταση της εργασίας σε όλους τους τομείς ε, με υψηλά, αναβαθμισμέ, υψηλά αναβαθμισμένες επιδόσεις χωρίς να αγνοούμε την ε, ένταξη της ισότητας των φύλων καθώς επίσης και τον αντίστοιχο κανονισμό για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των, των γυναικών την καταπολέμηση του γενετήσιου ακροτηριασμού των, του ακροτηριασμού των, γενε, ε, των οργάνων των γυναικών καθώς επίσης και για τη χορήγηση απαλλαγής που λέει ότι εγκρίνεται και καλούνται τα μέλη να συντάξουν τροπο, τροπολογίες σε σχέση με τη γνωμοδότηση η προθεσμία είναι η 6 Δεκεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών στις 17.00 στις 5 το απόγευμα και υπάρχει πραγματικά εδώ αναφέρεται ότι είναι ένας εξαιρετικός φορέας αυτό το Ίδρυμα για την ισότητα και πρέπει να υποστηριχθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, και τώρα να κάνουμε ένα γύρο και για να έχουμε αυτό το γύρο έχετε εσείς κυρία τον λόγο. Merci. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Και εδώ η συγγήτρια σκιώδης είναι η κυρία Ματέρα για το ΕΛΚΑ, για τους λόγους τους οποίους εξέφρασα προηγουμένως δεν είναι μαζί μας. Μου ζητά να ευχαριστήσω την κυρία Ντάντσιλα για την δουλειά την οποία κάνει, για την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητα. Για μας όλους και όλες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των αιτησίων του ετησίου απολογισμού που γίνεται με σαφή τρόπο ε, και διάφανο τρόπο και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε πλήρως με αυτά τα οποία είπε και έγραψε η κυρία Ντάντσιλα δεν υπάρχει κάποιο σημείο ανησυχίας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν από την κυρία Ματέρα έχουν την ίδια ακριβώς κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ κυρία Λεγκρίπ. Βάνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Και γι' αυτό το σχέδιο της κυρίας Ντανσίρα συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ τις συναδέλφους για την πολύ καλή δουλειά. Στι τροπολογίε που θα θέσουμε θα υπάρξουν συμπληρώσει και ενισχύσει κάποιων σημείων, ενδυναμωθούν κάποια σημεία. Και για τον εστιασμό, την επικέντρωση πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζονται περισσότερα στελέχη και δυναμικό. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να έχουμε συγκρίσιμου δείκτε και συγκρίσιμε πληροφορίε ώστε σε εύθετο χρονικό διάστημα να μπορούν να παρέχονται. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και να επιτευχθεί αυτή η διεύρυνση δυναμικού. Επίσης ε, η συνεισφορά αυτής της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε οι συνέργειες μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Ιδρύματος για την Ισότητα να ενδυναμωθούν, να ενισχυθούν και να μπορέσουν όλα αυτά να λειτουργήσουν ε, όπως και σε άλλες συζητήσεις τονίστηκε από πλευράς μας και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει αναφορά και στο καλό έργο που επιτελέστηκε πέρυσι από το Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Μπορεί το θέμα των δικτών ή ε, ολοκλήρωση της, ε, των στατιστικών στοιχείων για την ισότητα ή πλατφόρμα για την ισότητα μπορούν να συμπληρώσουν αυτό το τοπίο, αυτή την εικόνα. Σας ευχαριστούμε κυρία Βάνα. Και μετά από τις παρεμβάσεις αυτές σχετικά τώρα μπορούμε πράγματι να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, στην έκθεση για την ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να ολοκληρωθεί το χάσμα στις στις, ε, στην αμοιβή των γυναικών και των ανδρών. Έχει τον λόγο η συγγήτρια κυρία Λεγκρή. Oui, merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά συζητάμε σήμερα το απόγευμα αυτό το θέμα της έμονης παρουσίας διαφοράς στις συντάξεις ανδρών και γυναικών είναι γύρω στο 40%, 38% για τους άνω των 65%. Είναι ένα θέμα στο οποίο η Επιτροπή εδώ του Κοινοβουλίου δεν θα μπορούσε να μείνει αδιαφορή. Η ανταλλαγή απόψεων σήμερα αφορά τις διάφορες τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και οι οποίες προηγούνται της προετοιμασίας των συμβιβαστικών. Έχουν κατατεθεί 241 τροπολογίες από πλευράς των ε, εκπροσώπων των σκιωδών και όχι μόνο των σκιωδών αλλά και του συνόλου των πολιτικών ομάδων. Θέλω να σας συγχαρώ όλους για αυτό το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος για ένα σημαντικό βέβαια θέμα. Έχει γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες πιθανές συνενέσεις με βάση αυτές τις τροπολογίες. Θα ήθελα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια κοινά στοιχεία. Μετά από τις τροπολογίες αυτές, πολλά είναι τα θέματα τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα. Εγώ παρουσίασα κατά τη διάρκεια της, ε, του σχεδίου της εκθέσεως που είχα κάνει, είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στον στόχο της έκθεσης αυτής Πρέπει δηλαδή να μείνουμε πραγματικά ιδιαιτέρως κοντά στον βασικό μας στόχο, μια στρατηγική της Ένωσης, έτσι ώστε να σταματήσουν οι διαφορές της συντάξεις ανδρών και γυναικών. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μείνουμε κοντά στην έκθεση. Είμαι διατεθειμένη να συζητήσω με όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες και να εντάξω τους, τις ανησυχίες τους, χωρίς όμως να ξεφύγουμε από τον κεντρικό στόχο. Χρειάζεται μία προσπάθεια για να το πετύχουμε αυτό. Και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε μία ικανοποιητική απάντηση. Και έτσι μόνο θα αποφύγουμε μία μεγάλη διάχυση του μηνύματος το οποίο θέλουμε εμείς να οδηγήσουμε στην Ολομέλεια. Πολλές τροπολογίες επίσης με θετικό τρόπο ε, ταυτίζονται με τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις που είχα κάνει και αυτό με καθιστά ιδιαίτερο αισιόδοξη για τις συμβιβαστικές τις οποίες θα μπορέσουμε από κοινού να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει κάποια πράγματα να τα διευκρινίσουμε εδώ. Το θέμα της ανισότητας, σαν παράδειγμα ανδρών γυναικών στον τομέα αυτό, με διοικό τρόπο εκφράζεται επανειλημμένα. Έχω και εγώ επιμείνει στις διαφορές αυτές, περιγράφοντάς τες σαν ένα πολυπαραγοντικό και περίπλακο παράγοντα. Υπάρχει λοιπόν ένας διτός χαρακτήρας των αιτιών. Καταρχάς υπάρχουν διαφορετικές πορείες και διαδρομές επαγγελματικές και από την διαφορά του ύψους των αμοιβών από την άλλη. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε εμείς αυτό τον διοικό χαρακτήρα να τον περιγράψουμε σωστά και να σταματήσουν οι διαφοροποιήσεις αυτές, να διορθώσουμε μέσω των αντισταθμιστικών μηχανισμών ε, τις διαφοροποιήσεις οι οποίες εμένουν και θα πρέπει να καταργηθούν και ταυτόχρονα θέλουμε εμείς να προλάβουμε τις ανισότητες στον τομέα των εισοδημάτων των συνταξιοδοτικών έτσι ώστε η επαγγελματική πορεία του καθενός ε, ε, να ταυτίζεται όσο γίνεται περισσότερο σε επίπεδο φύλου. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ε, θα έλεγα αυτοί οι λόγοι συνδέονται ο ένας με τον άλλο και μιας και μπορούμε εμείς σαν προσπάθεια λύσης να μην αναφερθούμε αποκλειστικά σε ένα είδος δράσης, αυτό είναι θετικό. Γι' αυτό λοιπόν και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης ε, θα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εντάξουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης στο πλαίσιο ε, της εκθέσεως για τα συστήματα τα συνταξιοδοτικά και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Παραμένοντας πάντα επαναλαμβάνω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Επιτροπής ε, Υποθέσεων των Γυναικών. στα πλαίσια της επιστολής ε, διαμοιρασμού αρμοδιοτήτων που έχει υπογραφεί από τους Προέδρους των ε, επιτροπών. Λοιπόν, 241 τροπολογίες. Νομίζω ότι η προσπάθεια την οποία μέχρι τώρα κάναμε ήταν μια καλή προσπάθεια. Εγώ σε συνεργασία με όλους τους κοιόδης ε, προτείνω να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία έτσι ώστε στις 25 Φεβρουαρίου του 2017 να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νόηλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Αλλά τώρα δεν ομιλώ για την κυρία Ντανσίλα, αλλά για μένα προσωπικά είμαι σκιώδης εισηγήτρια και εγώ για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια στρατηγική για να αποφύγουμε την, να συνεχίζεται η διαφορά μεταξύ των φύλων. Αναφέρατε τον αριθμό των τροπολογιών. Αν δούμε τις τροπολογίες αυτές και τις βάζαμε σε μια στίβα, θα ήταν πολύ ψηλή, μεγάλο το ύψος αυτής της στίβας. Καταδεικνύεται έτσι ότι είναι πολύ σημαντικό να ενδιαφερθεί, να δώσει προσοχή σε αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση συσχετίζεται με την αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια των ατόμων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των γυναικών και συσχετίζεται με τις αρχές της ισότητας και έχουμε εδώ πολλές τροπολογίες που αφορούν το θέμα. Πολύ σύντομα λοιπόν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για την τελική κατεύθυνση. Ένα άλλο μεγάλο ύψος τροπολογιών, στίβα τροπολογιών αφορά τοποθετήσεις ότι πρέπει να συλλεγούν στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία για να μπορούμε να λάβουμε τις σωστές αποφάσει αποφάσεις και ότι ο στόχος ε, της ισότητας που θέλουμε να επιτευχθεί στο τέλος ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει να με, μεριμνήσουμε να επιμερίζουμε το έργο της φροντίδας στο σπίτι ή στο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί εκείνος ο οποίος κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά γυναίκες παίρνει μικρότερη σύνταξη στο τέλος τέλος και ανταμείβεται χειρότερα. Δεν μπορεί κανείς με επεφημίες και χειροκροτήματα να ζει, χρειάζεται χρήματα. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν η συνεισφορά ε, για τις γυναίκες ε, στις συντάξεις. Πρέπει να μεριμνήσουμε για μια ελάχιστη σύνταξη, ώστε να μπορεί να συνδυάζει την αξιοπρέπεια διαβίωσης και το αναγκαίο ποσό για αυτό, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Και θα προστατεύει <clears throat> τον, το να περιθωριοποιούνται οι γυναίκες κοινωνικά ή ε, μέσω των ε, καταστάσεων που δημιουργούνται διότι κάποιος ο οποίος ε, βρίσκεται σε υποδέστερη κατάσταση όχι μόνο είναι φτωχός αλλά και περιθωριοποιείται. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ελάχιστη σύνταξη, ελάχιστη σύνταξη και για τις γυναίκες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για τη διαπραγμάτευση. Μια ιδέα που οδηγεί σε μια νέα κατεύθυνση στην Ευρώπη σε σχέση με τον άνδρα που τρέφει την οικογένεια, δηλαδή αν εκείνος παίρνει αρκετά χρήματα αυτό είναι ικανοποιητικό. Όμω αυτό είναι ένα παροχημένο πρότυπο δεν μπορεί να συνεχίζεται στη σύγχρονη εποχή. Οι γυναίκε δεν μπορεί να κάνουν περισσότερη δουλειά και να παίρνουν μικρότερη σύνταξη. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε έχουν μεγάλη προοπτική και προέκταση για το μέλλον. Πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε μοχλευτικά όλα αυτά τα επιχειρήματα ώστε να επιτευχθεί ισότητα υπέρ των γυναικών. Και εδώ δεν είναι μόνο το θέμα του να ερευνήσουμε πώ μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Πρέπει να καταπολεμηθούν στερεότυπε εικόνε και σύμβολα. Δηλαδή αν δεν δεν υπάρξει καταπολέμηση των αιτίων δεν θα υπάρξει λύση υπάρχουν λαθασμένα κίνητρα για τη φορολόγηση. Έχουμε λαθασμένα πρότυπα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των ανδρών και οδηγούνται οι γυναίκες σε ένα αδιέξοδο. Τα χρήματα τα οποία οι γυναίκες μέσω ε, της δικής, της, ε, της δικής τους ζωής ε, θα έπρεπε να εισπράξουν όταν παίρνουν διαζύγιο από τους άνδρες τους δεν τα παίρνουν ποτέ. Χρειάζονται λοιπόν νέες στρατηγικές. Δεν χρειάζονται νέες στρατηγικές. Επαρκούν κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να είναι σεβαστές. Και πρέπει όταν προέρχονται από τις ίδιες γραμμές αυτές οι κινήσεις υπάρχει η μεγαλύτερη απειλή για τις γυναίκες, η μεγαλύτερη βία εις βάρος των γυναικών, η φτώχεια. Κάτι πρέπει να γίνει για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση. Σίγουρα θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη να συμβάλλουν όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Πώς είναι δυνατόν εδώ να μην διεκδικούμε κάτι μακροπρόθεσμα. Μέσω της αναμεταμόρφωσης της ε, κοινωνίας ε, μέσω του μεγάλου διαστήματος ε, που έχει μεσολαβήσει και δείχνει ποια είναι η μελλοντική κατεύθυνση πρέπει κάτι να κάνουμε, να επιλεγεί μια στρατηγική ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι γιατί διαφορετικά δεν θα βγάλει πουθενά αυτό. Επίσης αναφέρθηκε ότι το επάγγελμα και η αμοιβή πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο για να μπορέσει να επιτεθεί ισότητα το πρότυπο του άνδρα που διατρέφει την οικογένεια πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι το κλασικό θέμα που πάντα αφορούν τις γυναίκες όλα αυτά και που βρίσκονται σε υποδέστερη θέση. Όχι μόνο η πληρωμή αλλά και η αρνητική θέση της γυναίκας. Αυτό φαίνεται αμέσως και από ένα τραπεζικό αντίγραφο όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών. Ό,τι και αν κάνει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, στο τέλος τέλος ε, πληρώνει εκείνη τα σπασμένα και βλέπω, θεωρώ με την προθυμία που έχουμε να συνεργαστούμε θα μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς. Όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι συμβιβασμοί πρέπει να αποφασίσουμε μέσω της ψήφου μας. Ευχαριστώ. Hay más intervinientes. La señora Legrip ha hecho referencia al... Η κυρία Λεγκρίπ μίλησε για το χρονοδιάγραμμα και για τις επόμενες συναντήσεις, γιατί θα πρέπει και κάποιες από να τις ε, ε, διαπραγματευτούμε. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συνάντησης. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.